Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Έχουμε την κοινή εξέταση μια σειρά εκθέσεων. Καταρχήν την Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Είναι ο κύριος Πάετ, ο οποίος έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι.